Το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου έχει ο κύριος Λόπες Γκαρίντο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να τοποθετηθούμε όσον αφορά αυτή την αποστολή διακρύβωσης των γεγονότων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτό έγινε τέλη του 2008 στην Γάζα και τελείωσε αρχές του 2009 και αυτά όλα αποτυπώθηκαν στην λεγόμενη έκθεση Goldstone. Ακριβώς όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση του Μπάνκι ki προς το Συμβούλιο Ασφαλείας τον Ιανουάριο του 2009 έγινε μια ενημέρωση σε σχέση με τις ε, εντυπώσεις από την κατάσταση στη Γάζα. Επίσης, ακολούθησε δημοσίευση αυτής της ε, έκθεσης, αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, σε κάποια από τις συζητήσεις που κάναμε. Αυτό για το Σεπτέμβριο πέρσι. και έγινε σχετική συζήτηση στις 14 Ενάτου και 2 Δεκάτου στη 12η Σύνοδο του Συμβουλίου των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ιδέα Ευρωπαϊκή η ευρωπαικη ενωση αυτη εξ αρχή ε, τη σχετική σύγκρουση είχαμε επιμείνει ότι θα πρέπει τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να σεβαστούν τι ε, δεσμεύσει του στο διεθνέ δίκαιο. Και γι' αυτό παρακολουθήσαμε τι σχετικέ έρευνε κατόπιν των καταγγελιών για, για τι παραβιάσει. Η Σουηδική Προεδρία στην Γενέβη είπε ως θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η έκθεση αυτή έχει πάρα πολύ σοβαρές καταγγέλειες σε σχέση με σοβαρές παραβιάσεις ε, του διεθνούς ε, δικαίου γιατί αφορά ε, επιθέσεις κατά αμάχων. Οπότε θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν ε, ε, ε, κάποιες έρευνες εις βάθος για αυτές τις παραβιάσεις για να δούμε τι έκαναν οι εμπλεκόμενοι και να γίνουν αυτές οι έρευνες σύμφωνα με τα σχέδια του διεθνές δίκαιο. Οπότε υπήρξαν κάποιες συστάσεις και προς τα δύο εμπλεκόμενα μέρη από αυτήν την ε, αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε αυτή την τοποθέτηση στην έκθεση Γκόρθων και εκεί τονίστηκε στην συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 17 Ιανουαρίου, μόλις πριν από ένα μήνα, το πόσο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει αυτές οι έρευνες να προχωρήσουν, να γίνουν αξιόπιστες για αυτές τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Μπορώ δε να σας ενημερώσω ότι στις 4 Δευτέρου, αυτό το έτους, ο Γενικός Γραμματέας δημοσίευσε τη σχετική έκθεση. Δηλαδή, το ψήφισμα που αφορά την έκθεση Goldstone. Ισραήλ, Ελβετία και κατεχόμενα, όπου κοινοποιήθηκε αυτό το ψήφισμα πιο πριν δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουν οι έρευνε μέχρι να γίνει δημοσίευση αυτή. Οπότε όλα αυτά συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προτεραιότητα δε τη δική μα Προεδρία είναι να πετύχουμε συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια τοποθέτηση σε σχέση με αυτό το σχέδιο κειμένου που πρόκειται να παρουσιαστεί στο ΟΗΕ από πλευρά των Παλαιστινίων. Και ο στόχος μας είναι διτός. Αφενός, να υπάρχει συνετική έγκριση αυτού του κειμένου ή, ή να έχουμε όσο γίνεται πιο ομόφωνη στάση και φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, επαναλαμβάνουμε ότι η Προεδρία είναι υπέρ των όσων ζητά η έκθεση της ευρωπαικης ενωσης οποτε παραλαμβανουμε οτι η προεδρια ειναι υπερ των οσων ζητα η εκθεση κοστων δεν έχουμε κάποια ανεξάρτητη, αμερόληπτη ε, έρευνα των όσων έχουν γίνει στη Γάζα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεωργίευα, εκ μέρους της Επιτροπής. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω αυτά που είπε η Ισπανική Προεδρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστήριξε όλα τα ψηφίσματα, παρόλα αυτά ήταν σαφής η στάση της για την έκθεση Goldstone. Καλούνται όλα τα μέρη της διαμάχης να ξεκινήσουν έρευνας όσον αφορά υποψίες παραβιάσεων από τα αντιμαχόμενα μέλη του Διεθνούς Νόμου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Μέχρι στιγμής βήματα που έχει αναλάβει το Ισραήλ, οι Παλαιστινικές Αρχές και η Χαμάς δεν δίνουν απτά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι υπεύθυνο και υπόλογο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει το κύριο της μήνυμα ότι τα μέρη της διαμάχης θα πρέπει να ελέγξουν ακριβώς αυτές τις υποτιθέμενες παραβιάσεις. Και θα ήθελα να επιθυμίσω ότι η Κομισιόν δίνει σημαντική χρηματοδότηση σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που ο στόχος τους είναι να βοηθήσουν περαιτέρω και να προστατεύσουν Παλαιστίνιους άμαχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ε, να δοθούν οι απαραίτητες συνέχειες στο Συμβούλιο Άρχιας και να προσπαθήσουμε να βρεθεί μία επίλυση του προβλήματος. Κοινή συνενέση. Και θα ήθελα να σας πω ότι η Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία υπέβαλε ένα ψήφισμα για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της, ε, των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της έκθεσης Goldstone. Η, Goldstone, η Παλαιστινιακή πλευρά είπε ότι θέλει να προσπαθήσει να βρει μια λύση στις 26 Φεβρουαρίου, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και να επαναληφθούν τα σημαντικότερα σημεία του ψηφίσματος 64 καθώς 10 και να καλυφθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να ξαναπαρουσιάσει μια έκθεση σε 6 μήνες. οι διαβουλεύσει στον τομέα αυτό έχουν στο στόχο να επιτευχθεί μια κοινή λύση του θέματος και θα ήθελα να σας πω ότι υποστηρίζω την ε, άποψη της Ισπανικής Προεδρίας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, αναζητηθεί μια κοινή κοινοτική θέση και να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό που υπήρχε στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Εξ των πολιτικών ομάδων, πρώτος ο κύριος Μπροκ για δύο λεπτά. Πρόεδρε, Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αυτό που ελέγξα νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μία πραγματική έρευνα όσον αφορά τις ε, δεγόμενες παραβάσεις των θρημοδογημάτων είναι σημαντικό και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει να εξεταστεί. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στέφτηκε προς τα δύο μέρη, δηλαδή και εκείνων που ακολουθούν ένα ανσύμετρο τρόπο πολέμου, μια σύμμετρο μέθοδο πολέμου και ορίζουν το πεδίο μάχης με όλα τα προβλήματα που μια τέτοια ασύμετρη μορφή πολέμου επισύρει. Θεωρώ ότι αυτά όλα καταδεικνύουν ότι στη Μέση Ανατολή αλλά και σε άλλες παρόμοιες περιοχές μόνο μια ελληνική λύση θα μπορέσει να είναι πραγματική λύση. Εφόσον δεν υπάρχει ελληνική λύση δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ελέγξουμε τα προβλήματα αυτά. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανησυχίες του κράτους του Ισραήλ. και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή νέοι πύραυλοι που είναι επίση ανησυχητικοί. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό τη διεθνή ε, έρευνα είναι σημαντική, αλλά δεν ε, ολοκληρώνεται τα πράγματα με την έκθεση κορυφών. Θα πρέπει να εξασθούν τα κατεχόμενα. Είδαμε ότι όσον αφορά το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κανένα κράτος μέλος δεν υπερψήφισε αυτό αυτή την έκθεση. η καταψήφισαν ή απόσχον ή όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχαν καν στην ε, ε, ψηφοφορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες που υποστήριξαν το ψήφισμα είναι χώρες ε, όπως η Λιβύη, η Κίνα, ε, η Κούβα που καταπατούν ήδη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μην να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να ε, ασκήσουμε πολιτική κατά μία πλευρά. Η κυρία Ντεκάιζερ για δύο λεπτά. Δεκέμβριος 2008 η επιχείρηση σκληρό μολύβι στην Γάζα, οικογένειες κατεστραμμένες, καμένα σχολείο ε, ένας πληθυσμός ε, που ήταν ε, εγκλωβισμένο και δεν μπορούσε να ξεφύγει. Είμαστε, είχαμε μείνει άναυδοι γιατί μια τέτοια τραγωδία μπορούσε να εκτελεχθεί μπροστά στα μάτια τη διεθνού κοινότητα χωρί να κινήσει κανεί το μικρό του δαχτυλάκι. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Η πολιορκία συνεχίζεται. Όμω η έκθεση Goldstone υπάρχει. Είναι διαφορετική από το ψήφισμα που ακολούθησε. Η έκθεση Goldstone, αυτή η, θα, η θαραλέα έκθεση που δείχνει απλά πώ θα πρέπει να γίνει να ισχύσει δικαιοσύνη, είναι υπερβολικό αυτό αυτό. Οι πιέσει ε, να θαυτεί αυτή η έκθεση. Και ε, όλα αυτά είναι πραγματικά αφάνταστα. Τον διασύρουν, τον σέρνουν στη λάσπη. Δεν είναι ο μόνος ο οποίο ε, το, το Ισραήλ. Όμω θα σα πω και σαφώς και ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι η μόνη που κάνει να βασιλεύει ο τρόμο και λογοκρίνει την έκθεση. Και να σα πω κύριε Λίμπερμαν, δεν, ήσασταν, ε, δεν είσαστε εδώ, αλλά ήσασταν εχθέ στο Κοινοβούλιο. Δεν μα τρομάζετε εδώ. Δεν μπορείτε να μα εκφοβήσετε εδώ στο σώμα αυτό. Θέλουμε ανεξάρτητε έρευνε σε σχέση με τα διεθνή στάνταρ και όχι στρατιωτικά δικαστήρια που θα κρίνουν του ίδιου του φαντάρου, φαντάρους, τους στρατιωτικού. Να σα πω κύριε Λίμπερμαν, δεν είστε ευπρόσδεκτο. Όχι γιατί αντιπροσωπεύετε το Ισραήλ, αλλά γιατί θέσεις σας ρατσιστικέ και ξενόφοβε δεν είναι σύμμορφε προς τις ευρωπαϊκές αξίες. Κανένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να επιτρέψει την υπέρβαση του διεθνούς δικαίου χωρίς να υποστεί τις συνέπειε, χωρίς να δώσει λογαριασμό. Και αυτό το κοινοβούλιο δεν θα φεθεί στον εκφοβισμό. Θα συνεχίσει απλώς να ζητά να ισχύσει δικαιοσύνη και να χυθεί φω στην τραγωδία τη Χάζα χωρίς ε, ε, να είναι προκατελημένο, αλλά ε, όντας αποφασισμένο και ζητώ από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν σε αυτό να μείνουν. Δηλαδή στο φως και στη δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Η κυρία Νέιτς Ιτεμπρόκ για δύο λεπτά. Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα, η έκθεση Goldstone προσπαθεί να προβλέψει μια να, τηρήσει μια εντολή που δόθηκε και η εντολή ήταν η εξή να διερευνηθούν όλες οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που μπορεί να έχουν ε, γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξήχθησαν στην Γάζα κατά τη διάρκεια της περίοδου από τις 27 Δεκεμβρίου 2008 και τις 18 Δεκεμβρίου, ε, Ιανουαρίου 2009 είτε ε, ε, πριν, κατά τη διάρκεια, είτε μετά. Και ακριβώς αυτό είναι η έκθεση Γκόλστον. Δεν είναι μόνο ο κύριος Γκόλστον, ήταν και δύο ε, θηλυκές συνάδελφοι. Αυτό έκαναν, αυτό έρευνα έκαναν για το τι συνέβη στην Γάζα. Και προ... κατέληξαν σε πορίσματα τα οποία πραγματικά είναι ενοχλητικά, για να πω το πω έτσι ε, ε, απαλά και ελαφριά, γιατί τις περισσότερες φορές αποδείκνυουν ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου και παραβιάσεις των, της σύμβασης της Γενέ, των συμβάσεων μάλλον της Γενέβης έχουν διαπραχθεί από τις αρχές ενός κράτους που ισχυρίζεται ότι είναι το μόνο δημοκρατικό κράτος στην περιοχή. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικό και δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Όταν λοιπόν μας ζητάτε να λάβουμε θέση για αυτή την έκθεση, το θέμα δεν είναι αν είμαστε υπέρ υπέρ ή κατά του Ισραήλ, υπέρ ή κατά της Παλαιστίνης, υπέρ κατά της Αμάς. Το θέμα είναι αν ε, μπορούμε να ανεχτούμε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των συμβάσεων της Γενέβης, ανεξάρτητα από ποιο τις διέπραξε. Αυτό είναι που πρέπει να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. κυρία Λούκας για σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω πόσο ευτυχής είμαι που, επιπλέον, επιτέλους συζητάμε την έκθεση Γκόλσον στην Ολομέλη γιατί είναι ζωτική σημασία σε αυτό το θέμα και σήμερα η Ένωση ήταν ε, ε, ντροπιαστικά απούσα μέχρι σήμερα σε αυτό το θέμα παρά ότι έπρεπε να, το Συμβούλιο να κάνει συστάσεις για την έκθεση Γκόλσον τις οποίες υποτίθεται λαμβάνει σοβαρά υπόψη η Κομισιόν λέει το Συμβούλιο θα το υποστηρίξει μα δημοσίως πρέπει να γίνει αυτό και το ολόκληρο το Συμβούλιο θα πρέπει να το κάνει. Και είμαι ευτυχή που στο σχέδιο ψηφίσματο του Κοινοβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα το ψηφίσουμε αύριο έχουμε δύο πολύ ισχυρέ ε, παραγράφου που ζητούν από τον ΥΠΑ το εκπρόσωπο και τα κράτη-μέλη δημοσία να ζητήσουν ε, την εφαρμογή των συστάσεων τη έκθεση. Το ψήφισμα επίση του ζητά ενεργά να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των συστάσεων για τη διαβούλευση των εξωτερικών ε, αποστολών τη Ένωση και των ΜΚΟ επιτόπου. Γιατί οι αποδείξει που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε οι αρχές του Ισραήλ ούτε οι ΑΜΑΣ ε, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους ε, και μάλιστα με σοβαρό τρόπο. Και οι έρευνες ε, όσον αφορά τους στόχους και τις τακτικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του, της επιχείρησης αυτής πραγματικά αμφισβητούν την ανεξαρτησία των πορισμάτων και η Χαμάς δεν μπόρεσε να απαντήσει όσον αφορά την, ε, τους πυροβολισμούς που ε, ε, έκανε έναντι αμάχων πληθυσμών. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί στη Γάζα, στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζεται εκεί και πάλι από το Συμβούλιο και τον είπα το εκπρόσωπο να πιέσει το Ισραήλ να άρει την πολιορκία που εμποδίζει την ανοικοδόμηση και, το... και αυξάνει τη... τα προβλήματα εκεί. Ο κύριος Πανίσκη. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η έκθεση Goldstone ε, έχει έλλειμμα ισορροπίας και δίκαιης αντιμετώπισης διότι έχει συνταχθεί από τον ΟΗΕ ε, ενώ αφορά Ιράν, Σομαλία και άλλες χώρες που ανήκουν στον ΟΗΕ αλλά αυτές οι χώρες έχουν κάποια δικαιώματα όταν λοιπόν αυτές οι χώρες δεν αντιμετωπίζουν την ανθρώπινη δικαιώματα ως σοβαρή υπόθεση πώς Πώ γίνεται να επικαλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. επομένω πρόκειται για κάποια πηγή ύποπτη. Είναι η πηγή αυτή τη έκθεση, που έχει κάποια αιμονία, αιμονία κατά του Ισραήλ. Γιατί έχουμε 25 ψηφίσματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, διεκπαιρεώθηκαν από την ε, Επιτροπή και από τα 25 τα 20 ήταν κατά του Ισραήλ, ενώ κανένα ψήφισμα δεν αφορούσε άλλε χώρε που επίση αναφέρονται από την Επιτροπή αυτή. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα γυναικών, και άλλα. Μια που θεωρώ ότι, γι' αυτό το λόγο ότι εδώ λείπει η ισόρροπη αντιμετώπιση. Έχουμε τις ε, τρομακτικές συνέργειες της ε, Χαμάς που δεν αναφέρονται και επί 8 έτη είχαμε χιλιάδες πυράβλων που εκτοξευόντουσαν κατά αμάχων Ισραηλινών και άρα δικαιούται να προστατεύει τους πολίτες του το Ισραήλ κατά αυτών των τρομοκρατών. Έχουμε πάνω από 150 μηνύσεις κατά Ισραηλινών στρατιωτών. Πολλές φορές τα μη μεύσονικοί και ο τύπος γενικότερα επικρίνουν τις ελληνές αρχές, αλλά τίποτα δεν γίνεται σε σχέση με τους τρομοκράτες άλλης πλευράς. Επομένως εδώ πέρα υπάρχει έλλειμμα δικαιοσύνης και ισορροπίας ε, θεωρώ ότι θίγεται ένα βασικό μα σύμμαχο τη Μέση Ανατολή, αλλά δεν είναι σοβαρή έκθεση. για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, η έκθεση του δικαστή Goldstone είναι πιο τρανή απόδειξη για τα εγκλήματα, τη παραβιάση του διεθνού δικαίου και του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό. Από την έρευνα αναφύονται ισχυρέ ενδείξει, ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διέπραξαν σοβαρέ παραβιάσει τη τέταρτη σύμβασης τη Γενέβης αξίζει να σημειώσουμε πω ενώ η παλαιστινιακή πλευρά αν και τη γίνεται κριτική μέσω τη Έκθεση, αποδέχεται το διεθνέ δίκαιο και ζητά την εφαρμογή του ενώ αντίθετα το ισραήλ αρνείται. ενώ κάποιοι επιχειρούν την αποδυνάμωση τη ισχύω τη έκθεση, εμεί καλούμε τα κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθούν στο ύψο των αρχών που διέπουν το διεθνέ δίκαιο και την ευρωπαϊκή ένωση και να στηρίξουν συζήτηση τη έκθεση στη γενική συνέλευση του οηε και κοινοποίηση στο συμβούλιο ασφαλείας με στόχο την τελική της επικύρωση και τη λήψη μέτρων. η έκθεση θα πρέπει να φτάσει προ εξέταση στο διεθνές δικαστήριο της χάγης. αν η ευρωπαϊκή ένωση ενδιαφέρεται ειλικρινά για την επίλυση του παλαιστινιακού προβλήματος τότε θα πρέπει να σταματήσει την ανοχή στα εγκλήματα γιατί η ανοχή μεταφράζεται σε ενθάρρυνση και συνενοχή. επιπλέον με βάση τα πορίσματα της έκθεσης θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα η αναστολή των ενεργειών αναβάθμισης των σχέσεων ευρωπαϊκής ένωσης και ισραήλ και εφαρμογή των προνοιών της συμφωνίας σύνδεσης. οι λαοί της παλαιστίνης και του ισραήλ έχουν κάθε δικαίωμα στο μέλλον και στη ζωή. δική μας υποχρέωση είναι να πιέσουμε για επιτεύξη δίκαιης λύσης και ειρήνης. η έκθεση goldstone θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να δοθεί νέα όθηση με στόχο την επιτεύξη δίκαιης λύσης. Ο κύριος Μπέλντερ για Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση Goldstone αποτελεί, έπαιξε ρόλο κλειδί στην τελευταία, επίσκεψή μας στο κράτος του Ισραήλ της δικής μας αποστολής εκεί. Εδώ μας έδωσαν διάφορες ενημερώσεις ε, για τα πριν και μετά την στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα με λεπτομέρειες. Μας εξέγησαν τις έρευνες που έγιναν και τις ιδιαίτερα λεπηρές καταγγελίες και κατηγορίες κατά των Ισραηλινών αρχών. Αλλά ε, πέρα από την έκθεση Γκόλστον έχει γίνει διερεύνηση κάθε σοβαρή καταγγελία. Αλλά πότε η ΑΜΑΣ θα αρχίσει να διερευνά τι δικέ τη δράσει, τι δικέ τη ενέργειε. Πρόεδρε, τα διαθέσιμα στοιχεία για τι επιχειρήσει στη Γάζα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία πω η ΑΜΑΣ επίτηδε εξέθεσε του πολίτε τη Γάζα σε πολύ μεγάλο κίνδυνο κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. Αυτό σε κάθε περίπτωση έγινε για την προστασία των ε, ε, Ισραηλινών πολιτών ε, έναντι των διαρκών επιθέσεων με πυράβλους από πλευράς των Παλαιστινίων. Οπότε, Πρόεδρε, πρόκειται για μια προκατηλημένη έρευνα που, είναι, που οδηγεί απλά στην καταδίκη του Ισραήλ και καθιστά την ειρήνη δυσκολότερη στην Μέση Ανατολή. voorzitter vanaf het begin was duidelijk dat israël gebrandmerkt moest worden als dader. Ήταν σαφές από τις αρχές, πρόεδρε, ότι το Ισραήλ θα θεωρηθεί ο επιθέμενος στην ε, διαμάχη της ε, Γάζα. Ορισμένες χώρες ενθαρρύθηκαν ε, από την Αίγυπτο, το Πακιστάν και ξέρουμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες και εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα οπωσδήποτε δεν τη χάνουν σεβασμού. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μου ότι εδώ υπήρχαν χιλιάδες πύραυλοι εκτοκτευθήκανε από την Γάζα και γι' αυτό το Ισραήλ εκμεταλλεύτηκε το δικαίωμα αυτοάμυνας. Και η Χαμάς χρησιμοποίησε τον άμαχο πληθυσμό σαν ασπίδα προστασίας και εξετόξευσε τους πυράβλους από κτίρια πολιτικής χρήσης. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή θα πρέπει να πέσει αμέσως στον κάλαθο των αχρήστων. Ε, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν επιτρέπεται να διώκεται πολιτικά το κράτος της Ισραήλ κατά αυτόν τον τρόπο. Η κοινή γνώμη είναι διχασμένη σε σχέση με την έκθεση Γκόλστον. Ιδιαίτερα οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούνται πως ε, θελημένα προκάλεσαν το θάνατο πολυάριθμων αμάχων πολιτών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ε, ε, κατά της Γάζα. Όμως φαίνεται πως αυτό παραλείπει πολλά στοιχεία. Θα πρέπει να δούμε ότι πολλές κατοικίες που ήταν αποθήκες ε, εξοπλισμών, ε, στρατικών εξοπλισμών ε, και πυρομαχικών ήταν μέσα σε αυτούς τους στόχους. Επίσης, μετά από όλες αυτές τις προειδοποιήσεις, η αεροπορία θα είχε ρίξει μικρές, ε, μικρές μικρούς πυράβλους που θα ήθελαν μόνο να χτυπήσουν ε, τις συγκεκριμένες δομές. Ε, οι στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ είχε ειδοποιήσει τον πληθυσμό της Γάζας, χρησιμοποίησε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μπορεί να, κατα... να κατηγορηθεί πως ε, θελημένα χτύπησε άμαχο πληθυσμό. Εχθές την ίδια μέρα εγώ ήρθα σε επαφή με δύο πολύ σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες. Καταρχήν το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Λίμπερμαν και μετά τα απόγευμα με τον Αμπού Μάζερ, τον ε, αρχηγό τη Παλαιστινιακή Αρχή Και στι δύο περιπτώσει ήταν εκτεταμένε οι επαφέ με την ευχή επιτέλου να εγκαταληφθούν τα όπλα σε μια πορεία ειρήνη μετά από αγώνε που κρατούν εδώ και τόσε δεκαετίε. Η Ευρώπη, όπω ζητήθηκε και από τι δύο κυβερνήσει, θα πρέπει να διατηρήσει τον ισόρροπο ρόλο της του δικαστή χωρίς ε, προκαταλήψεις και ιδεολογικές θέσεις που μπορεί να δηλητηριάσουν τις ψυχές των μεν και των δε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εγώ θα αναλάβω τώρα την Προεδρία και θα μιλήσω ουγγρικά. Ορίστε Χάουιτ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ποιο από μερικέ μέρε ήρθε ο ύποπτο εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα και μα είπε ότι η έκθεση Gold Sword ήταν ει βάθο αντικειμενική και πληρούσε τα διεθνή πρότυπα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πετάξουμε στα άχρηστα την έκθεση αυτή. Α δράσουμε από αυτή. Εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με εκπροσώπου και τη Ιρανή κυβέρνηση των Παλαιστινιανών Αρχών και εκπροσώπους της ε, Κομισιόν που εξετάζει τα θέματα αυτά. Γίνονται ανεξάρτητες ε, έρευνες για να προωθηθούν αυτές οι εξετάσεις. Μίλησα με τον Μάρκο Πόρτσορ όταν είχε έρθει εδώ. Προς την Ισπανική Προεδρία έχω να πω, όταν προετοιμαστεί η ψηφοφορία στα Ηνωμένα Έθνη, δεν θα πρέπει να δικηβευτεί η συνένεση τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν υπήρχε ενιαία αποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν εις βάρος των θυμάτων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το κείμενο, αλλά ελπίζω περισσότερε από τι πέντε χώρε που υποψήφισαν την περασμένη φορά να το κάνουν τότε για να εξακολουθεί να ισχύει πίεση. Η έρευνα αυτή είναι πάρα πολύ σωστή. Όπω και η απόφαση του Διεθνού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2004 θα πρέπει να εξεταστεί σωστά και σύμφωνα με τα διεθνή σώματα. Εγώ καταδικάζω τη στάση των συντηρητικών που κατηγόρησαν το Ηνωμένο Έθνη. Και τα Ηνωμένα Έθνη αξίζουν πραγματικά τι υποστήριξή μα. Θα ήθελα να σα πω ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει υποφέρει από πολέμους θα πρέπει να καταδικαστούν ε, η, οποιαδήποτε εγκλήματα πολέμου. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να γίνονται δεκτά, να γίνονται αποδεκτά τα εγκλήματα αυτά. ευχαριστώ, Következő Madame Ries. Κυρία Αρίς, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, στόχος αυτής της συζήτησης δεν είναι να γίνουμε εμείς εισαγγελείς και να κρίνουμε αυτό που δεν ε, είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Είναι διπλός όμως ο στόχος μας. Καταρχήν να χυθεί φως στις ευθύνε των ΜΕΝ και των ΔΕ στον πόλεμο της Γάζα και πέρα από αυτό και με, πιο, με περισσότερη προοπτική να διερωτηθούμε πώς θα κάνουμε και τι θα πούμε σήμερα για να διευκολύνουμε την επιστροφή στο διάλογο. Και δεν πιστεύω πως η έκθεση Γκόλστον είναι επικοδομητική ε, για αυτό το οικοδόμημα και είναι καλό και πρέπει να το θυμίσουμε. Αυτό που κρίναμε το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή καμία δεν το υποστήριξε απέναντι στην εισαγγελία και οι μεγάλοι περασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι η Κίνα, το Πακιστάν, η Ρωσία και η Κούβα, για να σας πω μερικά ψηλοπαραδείγματα, η έκθεση είναι επίμαχη, είναι αμφισβητήσιμη ε, και είναι και προκατηλημένη. Θα πρέπει αντίθετα το Ισραήλ να αναλάβει τις ευθύνες, να αποφασίσει να αναλάβει αναλάβει τις ευθύνες του ως δημοκρατικό κράτος και να διαφωτίσει πλήρως το τι συνέβη στη Γάζα είναι συμφέρον του για το διπλωματικό ε, επίπεδο αλλά και έτσι όπως έχει πράξει και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κυρία, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι που πετύχαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε ε, σχετικά ευρεία πλειοψηφία για ένα ψήφισμα της έκθεσης Γκόλστον ε, χωρίς να μεταφέρουμε τη διαμάχη του ε, Μέση Ανατολής της Βρυξέλλες γιατί όπως θέλει να προωθήσει την ειρήνη θα πρέπει να προωθήσει αυτό που ενώνει τα δύο μέρη και όχι αυτό που τους χωρίζει και θα πρέπει να δούμε εδώ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά όπως θα πρέπει να επιτρέψουν τα διαμαχόμενα μέλη να έρευνα θα πρέπει επίσης να ε, δούμε και εμείς ότι δεν πρέπει να ε, κατηγορήσουμε μονομερώς το Ισραήλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί εκείνες οι χώρες που προσπαθούν να ε, αμφισβητήσουν την νομιμότητα του κράτους του Ισραήλ θα πρέπει να κατηγορηθούν από εμείς. Θα πρέπει να ενδυμανθούν εκείνες οι δυνάμεις στο Ισραήλ που θέλουν να προωθήσουν την ειρήνη και την ανοχή στην Μέση Ανατολική. Γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι η παρεμπόδιση των μη κοινωνικών οργανωτών στο Ισραήλ από την κυβέρνηση, παραδείγματο χάρη των Υπουργών Εξωτερικών κ. Λίβερμαν, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, γιατί αυτό διακυβεύει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο του ΟΗΕ το έκανε αυτό που είναι γεμάτο από εχθρού. Αλλά τι να περιμένουμε. Μεροληπτή απίστευτα. Και δεν έχει καμία νόημα αυτή η έκθεση. Δεν λέει τίποτα για τη χαμά και την τρομοκρατία του. Έχουμε 150 ε, πειθαρχικά τα οποία ερευνώνται στο Ισραήλ. Όμω υπάρχει μια ανθρώπινη τραγωδία πίσω αυτή την έκθεση, είναι η τραγωδία των Παλαιστινίων, οι οποίοι θέλουν επιστέλου κάποιου ε, νυφάλιου ηγέτε. Θέλουν ε, ειρήνη, θέλουν ευημερία. Και να μην ξεχνούμε επίση τι γίνεται στο νότιο Ισραήλ, που εκεί οι άμαχοι ε, χτυπώνται συνέχεια από τη Χαμάς και τους μανιακούς του ε, τζιχάντ με πύραυλους. Άρα μόνο η ειρήνη μπορεί να είναι μια βιώσιμη λύση για το Μεσανατολικό. Όμως δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό η έκθεση Γκόλστον. Η προσπάθεια κατά δυνατόν δυνατών ε, με Ισραήλ είναι για μένα ω Γερμανό και αριστερό μια, ε, κάτι το αυτονόητο. Δεν μπορώ όμως να δεχθώ ότι εδώ και πολλά χρόνια 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στο μεγαλύτερο ανοιχτό, ε, στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 44% των παιδιών κάτω των 14 ετών ζουν στη Γάζα. Καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πολιτική για το μέλλον της περιοχής. Προφανώς, ο πόλεμος του έτους 2008 θέλουμε να ξεχαστεί. Και γι' αυτό καλείται ε, να υπάρχει διαφοροποίηση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έτσι συνεχίζεται όμως αυτό το σπιράλ βίας. Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να εθελοτυφλεί και γι' αυτό θα πρέπει η έκθεση Γκόλτσο να εφαρμοστεί και αυτό θα είναι το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σόλτς. Φοντάνε, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε την έκθεση Goldstone με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά ε, τα ονόματα πολλών από τις χώρες που αποτελούν αυτή την ευρεία πλειοψηφία μας προβληματίζουν σε σχέση με την σύστασή του. Κίνα, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Δημιουργούνται λοιπόν ερωτηματικά όταν διαβάζουμε ότι αυτές οι χώρες, όχι τόσο υποδειγματικές στα θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλούν το Ισραήλ και την ΑΜΑΣ να διεξάγουν εις βάθος έρευνες για την κατα... παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Δεν θεωρούμε πως θα πρέπει να λάβουμε να κρατήσουμε τη μεριά του ενός ή του άλλου. Προτιμούμε να είμαστε ισορροπημένοι στην κρίση μας. Ευχόμαστε την ανάγκη να να, είναι εγγυημένη η ασφάλεια του Ισραήλ και των συνόρων του και το δικαίωμα της ύπαρξης του Εβραϊκού και του Παλαιστινιακού κράτους αντιθέμενη στη χρήση της βίας, της τρομοκρατίας και του πολέμου για την επίλυση των ε, συγκρούσεων. Η χριστιανική μας κουλτούρα μας οδηγούν στο να ευχηθούμε όλες οι παραβιάσεις να τιμωρηθούν με αυστηρό και ισόρροπο τρόπο. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά έχει το λόγο τώρα η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επανειλημμένα έχω υποστηρίξει ότι όταν δεν αναγνωρίζουμε το παρελθόν δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για αυτή τη σύγκρουση του Μεσανατολικού. Κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα πολλές επικριτικές φωνές ε, απέναντι στην έκθεση Γκόλστον. Εγώ γνωρίζω τον κύριο Γκόλστον από το καιρό εκείνο, όπου εκείνος ήταν ε, μεγάλος διαφημισολαβητής και έκανε πολλές έρευνες στην Νότια Αφρική. Ο κύριος Γκόλστον είναι και ανέκαθεν ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για να πλαισιώσει στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να φτάσει σε συμφιλίωση. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο εμείς εξετάζουμε αυτή την έκθεση δεν μας αφήνει να φτάσουμε σε συμφιλίωση και αντίθετα οδηγεί σε πόλωση της κατάστασης. Η έκθεση αγνοείται. Το Ισραήλ αγνοεί παντελώς την έκθεση αυτή Παρ' όλα αυτά, στο ΝΟΙΕ αναγνώρισε ότι έκανε σφάλματα και η Παλαιστινιακή πλευρά το αναγνώρισε αυτό. Ρωτώ λοιπόν, μήπως η Επιτροπή Έρευνα της Ραμάλα θα μπορέσει να κάνει μια σωστή έρευνα στην Γάζα και θα μπορέσει να οδηγήσει σε πορίσμα. Την επόμενη Παρασκευή έχω μια, υπάρχει μια συνεδρίωση στο ΝΟΙΕ και ελπίζω πραγματικά πως αυτή η συνεδρίαση ο νέος μας εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής θα μπορέσει να καταστήσει σαφή την ευρωπαϊκή θέση. Εμείς πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μερών, αλλά επίσης πάνω απ' όλα και σε κάθε περίπτωση, αν την Παρασκευή καταφέρουμε να έχουμε ομόφωνη γνώμη, εγώ θα είμαι ικανοποιημένη και πιστεύω πως θα προχωρούμε προς μια λύση στο Μεσανατολικό. Ευχαριστώ. Και τώρα, για ένα λεπτό, κυρία Σενιαλόβα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ταιριάζει να αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία όταν έχουμε ανθρώπινες ζωές που χάνονται, γιατί έχουμε εδώ πέρα πάνω από χίλιους οι οποίοι έχουν ε, υποστεί τις συνέπειες της σύγκρουσης. Ξέρουμε ποιος είναι ο και ποιος είναι το θύμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ιδίω μετά το 2006 έχουμε πάνω από χίλιους πυράβλους που έχουν εκτοξευθεί κατά άμα έχουν στο νότιο Ισραήλ. Δημόσια κτίρια και επικοινωνικές περιοχές έχουν πληγεί. Τι να κάνει το Ισραήλ, πώς να τους προστατεύσει. Οι άλλοι τους χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες τους αμάχους. Όμως και η διεθνή κοινότητα δεν έκανε τίποτα να προστατεύσει το Ισραήλ από τους ε, τρομοκράτες. Όλα αυτά είναι αμήλικτα ερωτήματα και θα πρέπει να απαντηθούν από την εξωτερική μας πολιτική. Με διάλογο και χτίσιμο εμπιστοσύνης μπορούμε να προχωρήσουμε προς μια βιώσιμη λύση στην Μέση Ανατολή και να κάνουμε να δούμε τις αιτίε της σύγκρουσης και αυτό που μπορεί να είναι σωστό βήμα. Πρόεδρο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Νικολό Ρινάλντι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση Γκόλστον ε, θέλει να αποτελέσει έναν ακρογωνιαίο λίθο για τον οποίο ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί οι πιθανές μελλοντικέ του διακλαδώσεις. Ε, Εμεί ε, δεχόμαστε πολλές επιθέσεις. Δεχόμαστε το αίτημα της έκθεσης για την διερεύνηση των θυμάτων σε άμα θέλουμε Θέλουμε ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα. Όπως αναφέρθηκε πολλές Ισραηλινές ε, ενώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν διαμαρτυρηθεί. Ακόμα και το κράτος ε, που φαίνεται πως έχει ε, εμπνευστεί από την μεγάλη ανθρωπιστική κουλτούρα του Ισραήλ, την εβραϊκή, της οποίας είμαστε όλοι κληρονόμοι. Εμείς ως Ευρώπη θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα πάνω απ' όλα στην Γάζα θα πρέπει να παραμείνουμε ανθρώπινοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρινάλντι και στη συνέχεια θα λέω το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Φρίντα Μπρέπουλς. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση Γκόλσταν αποδεικνύει με μεγάλη σαφήνεια ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Αμά έχουν ε, φέρουν μάλλον ε, την ενοχή για τις ε, επιθέσεις κατά μάχων ε, στην Γάζα. Και τα Ηνωμένα Έθνη πολλές φορές κάλεσαν τα δύο μέρη για να αναλυθεί η κατάσταση. Εγώ θα πρότεινα το εξής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει στο Διεθνές ε, Δικαστήριο, γιατί δεν πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ώστε να αποσαφινιστεί αυτή η κατάσταση και να σταματήσει η ατιμορρησία σε αυτή την περιοχή. Μα δεν μπορούμε να αφήνουμε να περνάνε ατιμωρητοί αυτέ οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτά τα εγκλήματα πολέμου δεν υπάρχει εδώ κανένα επιχείρημα το οποίο να μπορεί να σταθεί ώστε να μην εφαρμοστούν οι συστάσει αυτή τη έκθεση. Εγώ ελπίζω επίσης πως είπα του εκπρόσωπος και όλα τα κατημέλη θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ειρήνευση και να καταλήξουν σε επιτυχία έκβαση. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Είναι μονομερή αυτή η έκθεση, λέει ο κ. Φαντάλεν, διότι το Ισραήλ υφίσταται όλε αυτέ τις επικρίσεις ότι καταστρέφει οικονομικά αγαθά και, ε, και τους όμως ε, η Χαμάς από την μεριά κάνει τα ίδια. Η έκθεση όμως δεν το λαμβάνει αυτό υπόψη. Η έκθεση αυτή πηγαίνει μόνο το Ισραήλ. Ξέρουμε όμως ότι οι της Χαμάς χρησιμοποιούν κτίρια για μη στρατικούς σκοπούς και ε, νοσοκομεία κλπ. Φυσικά και πρέπει να γίνουν έρευνες όπως λέει η έκθεση. Και η Ζανή κυβέρνηση ορθώς έχει αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Έχουν αρχίσει οι σχετικές έρευνες και ανακρίσεις, κάτι το οποίο είναι θετικό. Όμως δεν νομίζω ότι η Χαμάς θα κάνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ λέει ο πρόεδρος. Ένα λεπτό. Πατρίκ Λιαρίκ. Εγκρίθηκε όμως από την συνέλευση, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη μα και οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Ένα είναι και μοναδικό το διεθνές δίκαιο, η ιδέα έκθεση Γκόλστον μετέρχεται αυτή, αυτό το χαρακτηρισμό εγκλήματα πολέμου. Κάτι το οποίο αφορά πράγματα που είδαμε όλες τις τηλεοράσεις και ακόμα και οι Ιρανοί στρατιώτες ε, κατήγγυλαν σε σχέση με ε, κάποιους ε, αμάχους που πυροβληθήκαν. οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει τις συνθήκες τόσο ώστε η Ισραηλινή κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τόσο επιτάσεις στο το διεθνές δίκαιο και να επιβάλλει και κυρώσεις αν χρειάζεται και αυτό να γίνει με αναστολή του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης του Ισραήλ με την ΕΕ, το οποίο προβλέπει. Η σχέση μεταξύ των ε, συμβαλωμένων θα πρέπει να δράζονται σε ανθρώπινα δικαιώματα και στην ε, δημοκρατία. Οπότε είναι σαφές και πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να ειδήσει και αποφασιστικό την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ακριβώς όπως προτείνει η έκθεση Γκόλστον. Και θα πρέπει και η Ολομέλεια να τοποθετηθεί στο εάν θέλει έναν κόσμο στον οποίο πρετανεύει η δικαιοσύνη ή ο νόμος του ισχυρότερο νόμος της ζούγκλας. Θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας σε σχέση με τους Ευρωπαίους αλλά και σε σχέση με τους λαούς όλου του κόσμου. Ο κύριος Μέσος για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση είναι κάτι το θλιβερό στην ιστορία της, ε, του του μια μαύρη σελίδα. Διότι δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το κείμενο αυτή την βροχή των πυράβλων που δέχονται οι άμαχοι στο Ισραήλ εδώ και τόσο καιρό. έχουμε όλα αυτά τα τούνελ που συνδέουν τη Γάζα με την ε, Αίγυπτο και άλλα μέρη ούτω ώστε να γίνεται λαθρεμπόριο όπλων και να μπορούν οι τρομοκράτες να επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, το Ισραήλ είναι κράτος δικαίου. Λειτουργεί ένα κράτος δικαίου. Ενώ από την άλλη μεριά στην Παλαιστίνη έχουμε τρομοκράτες. Οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν λόγο για τα εγκλήματά τους. Ήρθε τώρα με αυτή την έκθεση να καταθέσει κάποια πράγματα ο δικαστής Γκόλστον και επομένως είναι κρίμα που εμείς ε, μετερχόμαστε τέτοια επιχειρήματα εδώ. Για ένα λεπτό ο κύριος ε, Ντερόσα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούγοντας τη συζήτηση, θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι όλοι διαβάσαμε την ίδια έκθεση. Το Ισραήλ, το Ισραήλ αρνείται το δικαίωμα του συναστρίζεστε στο Ισραήλ και αρνείται την πρόσβαση στους δικούς μας υπουργού εξωτερικών. Χρησιμοποιούν επίσης ε, πλαστά ευρωπαϊκά διαβατήρια, το Ισραήλ ε, μας μεταχειρίζεται με περιφρόνηση. Αλλά αυτό δεν είναι εντυπωσιακό, δεδομένης ατιμορρησίας με την οποία συνεχίζει να παραβιάζει τα δικαιώματα εκατομμυρίων Παλαιστινίων αμάχων. Δική μας απάντηση θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη στην έκθεση Γκόλστον που ε, κατέληξε ότι αυτή η επιχείρηση ήταν απλώς ε, μια επιχείρηση στρατιωτική για να επιδιωχθεί περαιτέρω η πολιτική αυτή του Ισραήλ. Συστήνει η έκθεση το να πάει το Ισραήλ στο διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιμείνει για το κράτο δικαίου. Τέλο, εγώ υποστηρίζω την έκκληση του Γκόλστον στα κράτη-μέλη, τα συμβαλόμενα μέρη τη Σύμβασης τη Γενέβη συμπεριλαμβανομένη τη Ιρλανδία να αρχίσουν ποινικέ διώξει κατά των εγκληματιών πολέμου αλλά να κάνω μια διόρθωση πριν κλείσω. Ε, Επανειλημμένω ισχυριστήκαν διάφοροι ότι αυτή η έκθεση δεν ασχολείται με την, ε, με την ε, τους πυράβλους που, που χρησιμοποιεί η Αμάς κατά του Ισραήλ. Γίνεται η αναφορά από, για τις Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες οι οποίες πυροβολούν με πυράβλους στο νότιο Ισραήλ και όλμους. Ευχαριστώ. Θα πρέπει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάτσουν και να θυμηθούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα. Ο σκοπός της έκθεσης ήταν το να γίνει μία καταγραφή αμερόληπτη. Όμως δεν επιτεύθηκε ο σκόπος αυτός της έκθεσης, άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες όπως η Κούβα, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν. Χώρες που δεν ασπάζονται αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες. Επομένως, σκεφτείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Και εμείς να κάτσουμε επομένως να εξασφαλίσουμε κάποια ηγεσία ενιαία, στιβαρή στην Παλαιστίνη. Να σταματήσουν λοιπόν να υπονομεύουν οι Παλαιστίνοι και τη δική του δημοκρατία αλλά και του Ισραήλ. Επομένως είναι άλλη μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του ΟΗΕ. Υπάρχουν δε κάποιοι στρατιώτες του Ισραήλ που ακόμα κρατούν φυλακισμένοι και υπάρχει ένας Γάλλος στρατιώτη της επίσης. Και τώρα ο Τζέφρι Φαν Όρντεν έχει το λόγο. Ακούσαμε όλε αυτέ τι επικρίσει σχέση με την επέμβαση στη Γάζα και στο Ισραήλ. Όμω κανεί δεν λέει ότι δικαιούται η άμυνα, δικαιούται να λάβει δράση το Ισραήλ κατά αυτόν που θέλουν να σχεδιάσουν για να εκτελέσουν τρομοκρατικέ ενέργειε. Φυσικά και ο μέσος Παλαιστίνιος είναι συμπαθής και τον καταλαβαίνουμε, όμως επί 60 χρόνια έχουν ω ηγέτε κάποιου που είναι επαγγελματίε τρομοκράτε. Και ευθύ εξ αρχή, ε, ξέραμε ότι ε, ε, αυτό το όργανο του ΟΗΕ είναι πάρα πολύ επιλήψιμο και ακούσαμε και τον επικεφαλής επίσης ε, της ομάδας μας και ακούσαμε και άλλους που κάνουν μιλάνε μειωτικά γιατί ακριβώς ξέραμε ότι θα πρόκειται για καταδίκη του Ζαήλ, θα πρόκειται για μονόπλευρο κείμενο. Δεν λέει πάρα πολλά για Χαμάς αυτό το κείμενο. Δεν λέει για την τρομοκρατία, δεν λέει για τις επιθέσεις. Μιλά μόνο για τους ένοπλους Παλαιστινίους ε, και τι γίνεται με τους άμαχους. Εδώ έχουμε 500 σελίδες. Τίποτα από αυτές τις 500 σελίδες δεν έχει κάποια θετική πρόταση για βιώσιμη και σταθερότητα. Μόνο κοινή ρητορική. Επικρίσεις κατά του Ισραήλ. Όλα αυτά δεν περιποιούν τιμή στον ΟΗΕ. Ευχαριστούμε κύριε Φανόρντεμ, λέει ο πρόεδρος. Στη συνέχεια, Αλεξάνδρα Τάιν, έχετε το λόγο. Danke, Herr θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα στον ΝΑΕΑ υπάρχει ε, ε, το θέμα της ε, έκθεσης αυτής Goldstone που δεν σταματάνε οι πτώσεις, ιδίως όσον αφορά την Ισραηλινή πλευρά. Όσο και αν είναι αμφιλεγόμενη η έκθεση Goldstone, κάθε κράτος που θεωρείται κράτος δικαίου, δημοκρατικό, θα πρέπει να ελέγξει ανεξάρτητα αυτές τις, καταδι... Ε, κατηγορίες. Ε, δεν αρκεί μια στρατιωτική έρευνα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ακολουθήσει τις αρχές της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου θα πρέπει να ασχίσει περισσότερη πίεση και στα δύο μέρη μέσα στα πλαίσια διμερών σχέσεων για να εκδραστεί το θέμα της καταβάτησης του διεθνούς δικαίου. Εγκληματίες πολέμου θα πρέπει να κατηγορηθούν διεθνώς. Ίσως ο εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου θα πρέπει να δράσει βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 της συνθήκης της Ρώμης. Ε, τούτον δεν υπάρχει κανένας λόγο να τηρηθεί η πολιορκία της Γάζα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch Και πρώτα, ο κύριος Μικαλάσικ. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση Goldstone που συζητάμε αυτή τη στιγμή αγνοεί το δικαίωμα του Ισραήλ για άμυνα. Υπάρχουν πολύ έντονε κατηγορίε εδώ. Εγώ λυπάμαι όμω ε, τι οικογένειε, τα θύματα και θα πρέπει να πω ταυτόχρονα ότι υπήρχαν πολλέ. Ε, επιθέσεις από τη Χαμάς σε κατοικούμενες περιοχές του Ισραήλ. Και κάνω έκκληση να ζητήσουμε επίμονα να απανηθούν εκεί την βία. Ταυτόχρονα λοιπόν λοιπόν, που υπάρχουν τόσα πολλά θύματα. Χρειαζόμαστε έναν ε, καλό Παλαιστίνιο εταίρο, μια διάδοχο οργάνωση που θα εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα καρποφορήσουν όλες οι άλλες προσπάθειες. Θα πρέπει να διαράσουμε γλίγορα και που δεν, δεν επιτρέπεται να υποστηρίζουμε τους τρομοκράτες. Ευχαριστούμε κύριε Η κυρία Παπαδοπούλου έχει το λόγο η πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν βοήθα. στη γάζα έγιναν σωρία εγκλημάτων και γίνονται. υπάρχει φτώχεια εξαθλίωση βάναυση καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού. υπάρχουν μαρτυρίε γι' αυτό. υπάρχουν εκθέσει του ερυθρού σταυρού τη διεθνού τράπεζα του συμβουλίου τη Ευρώπη για εγκλήματα κατά των παλαιστινίων για οικονομική εξαθλίωση για απάνθρωπε συνθήκε διαβιώση στη γάζα. Α μην εθελοτυφλούμε. Η ανθρωπότητα γίνεται μάρτυρα βιοπραγιών εδώ και αρκετά χρόνια κατά των Παλαιστινίων. Η πολεμική μηχανή του Ισραήλ χτυπά ανελαίητα με το πρόσχημα τη αυτοάμυνα. Ο λαό των Παλαιστινίων υποφέρει. Καταδικάζουμε τι δολοφονίε αμάχων και στο Ισραήλ με όλη τη δύναμη τη ψυχή μα. Όμω, αυτόν δεν δίνει το δικαίωμα η άμυνα του Ισραήλ, η αυτοάμυνα του να σημαίνει διαρκώς καταιγισμό εναντίον και εγκλήματα εναντίον των Παλαιστινίων. Δεν δίνει το άλοθη στο Ισραήλ να κάνει τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. Σίγουρα δεν είμαστε εισαγγελείς όμως δεν μας αρμόζει ο ρόλος του πόντιου πιλάτου. Να νύπτουμε δηλαδή τα χέρια και να αφήνουμε την αιματοχυσία να συνεχίζεται και τα εγκλήματα του Ισραήλ να μένουν ατιμόρυτα. Με ευσεοποθισμό και απραξία αφήνουμε την ασυδοσία να οργιάζει. Αφήνουμε το θήτη ατιμόρυτο να ασελγεί κατά του θύματος. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αφήνουμε το δίκαιο του ισχυρού να επιβραβεύεται εναντίον του αδυνάτου. Következő hozzászóló Madame Barandika Bilbao. Στη συνέχεια θα λάβει το λόγο η κυρία Bilbao. Barandika. Barandika Bilbao. Barandika Bilbao, επαναλαμβάνει ο πρόεδρος. Ja, Michael Teurer ist mein Name. Ähm, Der Goldzoll-Bericht enthält Menschenrechtsverletzungen von... Λέγομαι Μιχαήλ Τόρες, κύριε Πρόεδρε. Ε, πάνω από 1.400 θύματα στην ε, ζώνη της Γάζας. Ε, πάρα πολλά, αλλά χωρίς επιθέσεις πυράβλων στη ζώνη δεν θα υπήρχε καμία άλλη επίθεση. Μια επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας επί τόπου είδαμε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και το Ισραήλ δεν επαφίεται και εξετάζει τι γίνεται. Δηλαδή η κεντρική ιδέα της έκθεσης Goldstone ότι το Ισραήλ ε, πει τούτου και συνεχώς επιτίθεται στον άμαχο πληθυσμό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει ο ξεχνάμε η Χαμάς χρησιμοποίησε τον άμαχο πληθυσμό για ασπίδα. Και εκτός αυτού δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει με τηλεφωνήματα και με φυλάδια που με έριξαν. Δεν έκανε το ίδιο το Χαμάς. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει για να αποφευθεί να εκτοξεύονται πύραυλοι της Χαμάς κοντά σε εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. αυτά που γίνονται ίσως δεν βοηθούν πολύ, αλλά εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε και από τις δύο πλευρές την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την επιστροφή στην ειρηνευτική διαδικασία. Συγγνώμη που έκανε λάθος όταν εκφώνησα το όνομά σας. Και ευχαριστώ που λάβετε το λόγο και τώρα. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κιλ Νίλσεν. Στο Ισραήλ έχει αμαυρωθεί τελείω και απαξιωθεί αυτή η έκθεση. Γιατί υπάρχει μια τέτοια εκστρατεία δυσφήμισης κατά των εμπεριστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έχουμε ένα καινούριο ίδρυμα το οποίο χρηματοδοτεί του βασικού φορεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και, πιο συγκεκριμένα, υπάρχει τέτοια εκστρατεία κατά τη κυρία Ναγμή Ραζάν που ήταν στην Κνεσέτ ε, βουλευτήνα, πανεπιστημιακή, ήταν διανοούμενη και έχει στρατευτεί για τα δικαιώματα των γυναικών και υπέρ τη ειρήνη. 13 τέτοιε ειρηνιστικέ οργανώσει, Breaking the Silence και άλλε, είναι στόχοι ενό τέτοιου κυνηγιού μαγισσών. Οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει αμελητή αυτές τις ε, οργανώσει. σε όλες τις χώρες, αλλά βέβαια και στο Ισραήλ. Πρόκειται για προσβολή προς την δημοκρατία. Άρα θα πρέπει να υπερσπιστούν το Ισραήλ κατά των δικών του των ίδιων των δαιμόνων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και στη συνέχεια θα λάβει ο κύριος ε, το λόγο. Ε, και οι δύο πλευρές φταίνε, αλλά υπερβάλλει σε σχέση με αυτή την έκθεση το Ισραήλ. Είναι δικαστής, σεβαστός. Είναι Ισραηλίτης. Φυσικά και δεν είναι τέλεια η έκθεση. Όμως, οι επικρίσεις βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά και έχουν καταθέσει σχετικά και κάποιοι στρατιώτες, Ισραηλινοί. Και η οργάνωση Breaking the Silence που ήρθε σε επαφή με αυτούς. Γιατί επομένως δεν γίνεται κάποια πραγματική έρευνα για κάποιους στρατιώτες οι οποίοι ίσω έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Και η Παλαιστινιακή οργάνωση επίσης ε, έχει δεχθεί κάποια σφάλματα. Να μην λοιπόν τόσο... Ε, ε μην έχουν τη στάση την αγέροχη Ιζελή. Πρόεδρος. Και τώρα στη συνέχεια θα λάβει το λόγο ο τελευταίος ομιλητής Κέλλη Σον. Οι λέξεις κλειδιά είναι ανεξάρτητος, δίκαιος, ουδέτερος. Θα πρέπει επομένω να έχουμε καταδίκη όλων όσοι παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Και επίσης χρειάζεται κάποιος ε, ουδέτερος να διαμεσολαβήσει. Όλα αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου να κάνει αυτό που έκανε ο Τζος Μίτσος στη Βόρεια Ολλανδία. Αυτοί που προβολούσαν πριν ένα στον άλλο τώρα συνεργάζονται για την ειρήνη. Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να βρούμε αυτή την ουδετερότητα, την αμεροληψία και την δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση μας που τώρα δεν ισχύει. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και... Τώρα, θα δώσουμε το λόγο. Α, υπάρχει ένα διαδικαστικό. διαδικαστικό. Διακόπτει ο Πρόεδρος για το διαδικαστικό. Uh, can I, can I ask... Εγώ θέλω να πεθεθώ στον κύριο Κέλλη. Είμαι βεβαία ότι με μεγάλη του χαρά θα διευκρινίσει το ότι το δικό μου κόμμα στη Βόρειο Ιρλανδία συμμετέχει στην κυβέρνηση και είναι φιλιρινικό. Ούτε σκοτώνει ούτε πυροβολεί. Ο IRA και η πολιτική του πτέρυγα κάνουν τέτοια πράγματα. Και τώρα θα δώσουμε στον κύριο Λόπες Γκαρίδο το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση είχε πλουραλισμό και αφορούσε και την έκθεση έκθεση γκόστον αλλά και την κατάσταση που οδήγησε στην σύνταξη της έκθεσης διότι νομίζω ότι θα πρέπει η Προεδρία να σας επαναλάβει ότι η έκθεση Γκόλστον είναι σημείο αναφοράς Το είπε το Συμβούλιο, το είπε η κυρία Γεωργίευα για την Κομισιόν όταν έλαβε το λόγο. Είναι σοβαρή η έκθεση. Φαίνεται ομερόληπτη και αντικειμενική και αναδεικνύει κάποιες πάρα πολύ σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παραβιάσεις από όλους τους εμπλεκομένους σε αυτή τη σύγκρουση. Και όπως είπαμε δεν είναι δυνατόν να μείνει Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον αυτής της καταγγελίας της έκθεσης. Διότι αντικειμενικά και σοβαρά η νυφάλια μας αναφέρει την πιθανότητα κάποιων φερομένων ως σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό το οποίο προτείνει η έκθεση, δηλαδή το να υπάρχουν ε, αξιόπιστες και αμερόληπτες έρευνες, να γίνει, γιατί είναι η πιο σωστή συνέχεια σε αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει, ως συνέπεια, να μας κάνει να τοποθετηθούμε όλους. Όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στο Κοινοβούλιο, σε όλους εμάς που πιστεύουμε στο ότι πρέπει να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάντοτε αντιδρούμε εις τέτοιες σοβαρές παραβιάσεις όπω εν προκειμένου ισχύει. Βεβαίω, και στον ΟΗΕ θα γίνει αυτή η συζήτηση, θα την στηρίξουμε και θα γίνει και στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η, επίσης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ασχολείται με τα καταγγελόμενα, οπότε και εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, όπως προείπαμε, να έχουμε Ευρωπαϊ... ε, συντονισμό και επικοδομητική στάση σε σχέση με αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά που καταγγείλει η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, την Επίτροπο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν ναι. σαφώς να δηλώσω πως η Κομισιόν με συνέπεια και με στένος έχει εκφράσει την μεγάλη της ε, ανησυχία για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα. Ο προκάτοχός μου, Λουί Μισελ, επισκέφθηκε τη Γάζα αμέσως μετά την επιχείρηση τη στρατιωτική ήταν αυτό από τις μάρτυρες παραβιάσεων και από τις δύο πλευρές και όρθωσε το ανάστημά του. και βροντοφώναξε την ύπαρξη αυτών των παραβιάσεων και την ανάγκη πλήρους σεβασμού από όλες τις πλευρές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου καθώς και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ανθρωπιστικές προσπάθειες για την ανακούφιση του πληθυσμού να μπορούν να φτάσουν στο πληθυσμό της Γάζας. Από τότε, έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει σαφές πως θα παρακολουθήσει στενά τις έρευνες για τους ισχυρισμούς παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και εξακολουθώ η Κομισιόν να υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδεσίας και της ε, πάυσης της ατιμορρησίας για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στην περίπλοκη διαδικασία ε, της Μέσης Ανατολής, ο σεβασμός του ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τόσο σημαντικό σήμερα όσο και ανέκαθεν και ίσως και ακόμη πιο σημαντικό για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιόπιστος εταίρος στην ε, ειρηνευτική διαδικασία είναι απαραίτητο να αποδείξει ότι εφαρμόζει τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης σε όλα τα πλαίσια σε κάθε πλαίσιο και ότι συμμορφούνται προς ε, τα κεκτημένα του διεθνούς δικαίου με συνέπεια και για οποιοδήποτε σημείο και θέμα. Και πάλι θέλω να υποστηρίξω την Προεδρία ότι μια κοινή ε, γραμμή της Ένωσης για την υπόθεση Γκόλστον θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε στην επόμενη σύνοδο.